Ladies and gentlemen, please take your seats. Καθίστε σας παρακαλώ. Because we have to proceed, we are... Πρέπει να προχωρήσουμε, έχουμε καθυστερήσει ήδη 10 λεπτά και έπονται και άλλες ε, συνεδριάσεις συγκρότησης σε σώμα. Άρα πρέπει να βιαστούμε. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ο στόχος της συνεδρίασης είναι να συγκροτηθεί σε σώμα η Επιτροπή με την εκλογή του Πρόεδρου και των τεσσάρων αντιπροέδρων βάσει του άρθρου 204 ε, του ιστορικού κανονισμού. Πρώτα θα προβούμε στην εκλογή του Πρόεδρου και στη συνέχεια θα εκλέξουμε τους αντιπροέδρους ενώ θα προεδρεύει ο εκλεγέντας πρόεδρος. Με ειδοποίησαν ότι τα εξής αναπληρωματικά μέλη θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και θα διαβάσω τα ονόματα. For uh, Mr. Lars Adaknusson, uh, there will be Mrs. Η κυρία Σουίτσα για τον κύριο Λάρς Αντάκτουσον, για τον, τη Μισελα Λιό Μαρή, ο Φιλίπ Ζουβά, για τον ε, Λορέντσο Τσέζα, ο Λουίς Τεγκράντες Πασκάλ, θα τον αντικαταστήσει, για τον Ραμόν Ραμανέσκο, η Μαρία Γκαμπριέλ, για όχι, ο Γιάννη Μουστέτιβα είναι εδώ. Για την Ελένη Θεοχάρους, η Ρενάτα Σόμαρ. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Μιλτιάδης Κύρκος. Ο Ρίτσαρτ Χάβιντ είναι εδώ. Θα αντικατασταθεί από την Ίνα Γκίλ. Ο κύριος Μπόρι Ζάλα από τον Ίσβα Βίχελη. Ο Ιωακίμ Σταρμπατή από τον Μάρεκ Ιούρεκ, Ο Ιβο Βάιγκελ από την Ανλή Γιατερμάκη. Ο Πάπλο Ιγκλέησιας του Ριών από τη Μαρή Κριστίν Βεργιά. Και ο Λουρίκε Λούνατσεκ από τον Ίγκορ Σόλτες. So, I will now ask... Τώρα ζητώ από την Γραμματεία να επαληθεύσει την απαρτία για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία. Ωραία. Ε, δυνάμει του άρθρου 208 του ιστορικού κανονισμού η απαρτία ισοδυναμεί στο 1 τέταρτο των μελών ε, προκειμένου 18 μέλη. Έχουμε απαρτία. Παρακαλώ υποβάλει τις υποψηφότητες για την Προεδρία. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει μια πολιτική ομάδα ή 5% των μελών της Επιτροπής να προτείνουν μία υποψηφιότητα, δηλαδή 4 μέλη στην περίπτωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Βλέπω ότι το ΕΛΚ έχει υποβάλει την υποψηφιότητα του κ. Μπροκ για την Προεδρία της Επιτροπής και ρωτώ αν συνενεί ο κύριος Μπροκ για την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ την πολιτική μου ομάδα για την υποψηφιότητα, λέει ο κύριος Μπρό, και τα υπόλοιπα σχόλια εκτός μικροφώνου. Δεν υπάρχει επιλογή, όπως σε όλες τις ε, δημοκρατίες. Ε, πληρούνται τα τυπικά ε, προσόντα. Α, ο κύριος Σταρμπάτη με ενημερώνει τώρα είναι εδώ. Θα ψηφίσει πληρεί ε, τις τυπικές υποχρεώσεις, είναι πλήρες μέλος ο κύριος Μπρόκ και έχει ε, υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Όχι. Θα εκλέξουμε διαβοή στον νέο πρόεδρο. Ποιοι είναι υπέρ. Όπως βλέπετε, ομόφωνα εκλέχθηκε ο κύριος Πρό, διαβοής. Τον καλό να έρθει στο Προεδρείο για να συνεχίσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμότατα και ελπίζω να συνεχίσουμε και τα επόμενα δυόμιση χρόνια τη συνεργασία μας σε συλλογικό πνεύμα. Μπορεί να έχουμε διαφορές από θέμα σε θέμα, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω προσπαθήσαμε να χτίσουμε γέφυρες και με μεγάλη πλειοψηφία να δρούμε κάθε φορά. Ελπίζω σε σημαντικούς τομείς αυτό να συνεχιστεί δεδομένης και της κρίσιμης κατάστασης ε, στην οποία ε, βρίσκεται ο κόσμος γύρω μας. Ερχόμαστε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων. έχουμε για τον πρώτο αντιπρόεδρο υποψηφιότητα. Ποιο είναι? Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών προτείνει τον κύριο Λεγκούτκο για πρώτο αντιπρόεδρο. Άλλες προτάσεις υπάρχουν? Όχι. Ο κύριος Λεγκούτκο είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής μας, τακτικό μέλος και έχει υπογράψει το πόθεν έσχες, δηλαδή τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, πληρεί τις προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος και δεν έχει ζητηθεί. Α, κατέφτασε ο κύριος Χάουιτ και θα ψηφίσει. Θα ψηφίσεις? Ωραία. Λοιπόν, ένα δικαστικό, διαδικαστικό έχω. Κύριε Λεγκούτκο, αποδέχεστε αυτή την υποψηφιότητα. E Είπαμε ότι ο, το ECR έχει προτείνει τον κύριο Λεγκούτκο. Έχετε κάτι ειδικό να πείτε. Ε, ε, μα δεν προτείνει ο πρόεδρος, η ομάδα προτείνει τον υποψήφιο. Τέλος πάντων θέλω να πω κάτι ειδικό για τον κύριο Λεγκούτκο, λέει ο κύριο Στάνοκ. Ε, που είναι πρώην γερουσιαστής ε, της Πολωνίας, ε, ηγείται τη Εθνική Αντιπροσωπή, είναι αντιπρόεδρο τη ομάδα μα και πενταετία είναι διακεκριμένο μέλο τη επιτροπή μα και άρα πληρεί κάθε προπόθεση για να καταλάβει αυτό το αξίωμα και με ιδιαίτερη υπερηφάνεια υποβάλλουμε την υποψηφιότητά του για την πρώτη αντιπροεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Απλούστευσα τη διαδικασία όπω και ο κύριο Πασκού στην δική μου μου περίπτωση είπα απλώς ότι έχει υποβληθεί η υποψηφιότητα. Μόνο αυτό έκανα. Υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος. Πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ε, διαβοής μπορούμε να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. The Ο κύριος Λεγκούτκο. Και αν θέλετε, ελάτε και στο βήμα. Now we have to come Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο αντιπρόεδρο. Μην κάνω πάλι το λάθος να διαβάσω αυτό που έχουν προτείνει οι πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ την ομάδα ποιον προτείνει. Η Γκουε νομίζω ότι και αριστερά πρέπει να προτείνει υποψήφιο. No from Δεν προτείνει η Γκουε τίποτα. Α, η κυρία Λούζιν. Το ξέρουμε ότι είστε τυφλός από το αριστερό μάτι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, ναι, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει με εμένα. Ε, λοιπόν, προτείνουμε την κυρία Μαρίνα Αλμπιόλ ως δεύτερη αντιπρόεδρο, γυναίκα της Επιτροπής. Ε, γεννήθηκε στην Καστελό της Βαλένσια στην Ισπανία και συμμετείχε στο κίνημα ειρήνης και διεθνής αλληλεγγύης από το 2000 ως νέα ακτιβίστρια έχει επικεντρωθεί στη δουλειά της κυρίως στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Εξελέγει το 2007 μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της ε, Περιφέρειας Βαλένσια και μέχρι να εκλεγεί Ευρωβουλευτής διατέλεσε μέλος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Εκλέκτηκε μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στο ψηφοδέλτιο Ισχέρδα ε, Πλουράλ, Ισχέρδα Ουνίδα. Ενωτική και πληθυντική αριστερά. Ευχαριστώ. Άλλε υποψηφιότητε υπάρχουν. Όχι. Η κυρία Αλμπιόλ είναι μέλος της Επιτροπής μας και έχει υπογράψει το Ποθενές για σύνδεση Οικονομικών Συμφερόντων, άρα πληρεί τις προϋποθέσεις για την κατάθεση υποψηφιότητα. Εφόσον δεν έχει ζήτηθει μυστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε διαβοής. Κυρία Αμπιόλ, αποδέχεστε αυτή την εκλογή. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια κυρία Αλμπιόλη για την εκλογή σας. Είμαστε τώρα στην εκλογή του τρίτου αντιπρόεδρου. Η σοσιαλιστική ομάδα παρακαλείται να καταθέσει υποψηφιότητα. Ο κύριος Χάουιτ έχει το λόγο. Ε, Καταρχήν ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένα. Με αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που υποβάλλω την υποψηφιότητα του κυρίου Πάσκου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκ των Σοσιαλιστών. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ευρωβουλευτές ότι ήταν ε, πολύ αξιόλογος αντιπρόεδρος στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και ιδιαίτερα διακεκριμένο μέλο, πρώην Υπουργό Άμυνα τη χώρα του, τη πατρίδα του τη Ρουμανία και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα ασφάλεια και άμυνα. Επίση είναι η Δήμον σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Και με ιδιαίτερη χαρά το υποβάλλουμε, υποβάλλουμε την υποψηφιότητά του για την αντιπροεδρία, τρίτη αντιπροεδρία τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Άλλε προτάσει υπάρχουν. Όχι. Ο κύριος Πάσκο Πλήρη επίση τι προποθέσει, είναι και πλήρε μέλο τη Επιτροπή μα, αλλά έχει υπογράψει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Άλλε προτάσει υπάρχουν, όχι. Μπορούμε λοιπόν διαβοή να τον εκλέξουμε. Ποιο υποστηρίζει τον κύριο Πάσχου. Αποδέχεστε την εκλογή σας κύριε Πάσκου. Συγχαρητήρια, παρακαλώ ελάτε και εσείς στο Προεδρείο. Τώρα θα πρέπει να εκλέξουμε τον τέταρτο αντιπρόεδρο. Με πρόταση νομίζω της ομάδας EFTD. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω με την κυρία Ιβέτα Γκρικούλη από τη Λετωνία ως υποψηφιό μας για την ε, Αντιπροεδρία. Δεύτερη φορά, δύο φορές εξελέγει εθνική βουλευτής και συμμετείχε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ήταν μάλιστα και αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής. Επίσης ήταν ε, μέρος αντιπροσωπείας για τις σχέση με τον ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι έχει πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό και πιστεύω ότι θα τιμήσει η παρουσία της στο Προεδρείο της ε, ομάδας, της Επιτροπής, συγγνώμης. Και ελπίζω η ΑΦΕΤ να τιμήσει και τις μικρές ομάδες και να σεβαστεί τα δικαιώματά τους και να μην επαναληφθεί αυτό που είδαμε χθε άλλη Επιτροπή. Και ελπίζω έτσι να έχει και η Λετωνία αντιπρόεδρο σε μια Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Γκρίγκουλε ε, πλήρη τις προϋποθέσεις, είναι μέλος της Επιτροπής μας και έχει υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Άλλες προτάσεις υπάρχουν υποψηφιότητες. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα του κυρίου Αντρέη Πλένκοβιτς. Για 17 χρόνια ήταν διπλωμάτης και υφυπουργό υποθε... ευρωπαϊκών υποθέσεων στην πατρίδα του, την Κροατία. Έχει επανεκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κροατίας. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελε να στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Πλέγκοβιτς που κάθεται δίπλα μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλες προτάσεις έχουμε? Όχι. Μόλις ρώτησα για τη διαδικασία και ο κύριος Πλένκοβιτς πλήρη τις προϋποθέσεις έχει υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και βεβαίως είναι και τακτικό μέλος της Επιτροπής μας και τυπικός πλήρη τις προϋποθέσεις. Τώρα θα κάνουμε μυστική ψηφοφορία αναγκαστικά. Παρακαλώ να διανεμηθούν τα ψηφοδέλτια. Α, όχι, ηλεκτρονικά θα το κάνω. Ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Έχετε παρακαλώ όλοι μαζί σας τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. The names printed in on that. Ονόματα τα λέει το μηχάνημα. Πλένκοβιτς και Γκριγκούλε παρακαλώ. Yeah, but it must be here in that they can vote. It's a secret ballot. Otherwise, we have to use paper. Green is candidate one, and red, red, red is candidate uh, number two. Uh, okay. We do not with... Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε, λέει, ονόματα στις οθόνες. Έχουμε μόνο κόκκινο και πράσινο. Κόκκινο είναι κυρία... Συγγνώμη, πράσινο είναι η κυρία Γκριγκούλε και το κόκκινο κουμπί είναι ο κύριος Πλένκοβιτς. Και το λευκό είναι λευκό, η αποχή. Mrs. Is... Η κυρία Γκριγκούλε είναι υποψηφιότητα της EFTD. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, προτείνει υποψήφιο τον κύριο Πλένκοβιτς. Η κυρία Γκριγκούλε, λοιπόν, το πράσινο κουμπί και ο κύριος Πλένκοβιτς το κόκκινο κουμπί. Ορίστε κύριε Τάνο. Επειδή είμαι πολλά χρόνια μέρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θυμάμαι ότι πριν από πέντε χρόνια επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο και ο κύριο Προβέρα και να διαταραχθεί το, το σύστημα DONT. Αν το διαταράξουμε το σύστημα DONT για μία ομάδα, θα πρέπει να το καταργήσουμε για όλε. Γιατί ε, δεν είναι σωστό, είναι παράτυπη η δεύτερη υποψηφιότητα. Αν ε, ε, καταργήσουμε για την περίπτωση αυτών των τεχών, θα πρέπει να το, να το παραβαίνουμε μονίμως αυτό τον κανόνα. Θα πρέπει να εξηγήσει την ομάδα σας αν συμβεί αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος ε, πάντα ε, αγνοεί αυτά τα πράγματα, δεν έχει ιδέα. Αλλά νομίζω επανειλημμένα το έχουμε δει και αυτές τις τελευταίες μέρες νομίζω έχει προκύψει. Αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα δεν μπορώ να την απαγορεύσω. Είναι θέμα δημοκρατίας. Ο κύριος Φλέκενστάιν να μας δώσει τη δική του θέση θέλει. Ναι, μπορεί να υπήρξαν κάποιες συμφωνίες. Το μόνο που γνωρίζω εγώ είναι ότι προβλέπει ο κανονισμός ε, πριν την εκλογή να μπορεί κάποιο να κατεβάσει πρόταση. Και αν κάποιο θεωρεί ότι θέλει να είναι υποψήφιο, ε, έχει το δικαίωμα να προταθεί. Θέλω να πω στους φίλους μου, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες είναι πάντα κόκκινοι. Αυτό ναι, Αυτός είναι ένα κώδικα που καταλαβαίνουν μόνο οι σοσιαλιστέ, από ό,τι φαίνεται. E λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. many people? There are 70, 74. ECR has one extra. There are Too many votes. We are 71. ECR has too many votes. ECR. Ψηφίζει ένας υπεράριθμος από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. ECR. We stop the vote. Θα σταματήσουμε την ψηφοφορία. Για να ελέγξουν παρακαλώ οι πολιτικές ομάδες αν ψηφίζουν ακριβώς τα μέλη που δικαιούνται. Ακούω ότι περισσεύει ένας από την ECR και από άλλα κόμματα άλλοι δύο. So, the EPP has... Το ΕΛΚ δικαιούται 21 μέλη. Παρακαλώ ελέγξτε πόσοι ψηφίζουν. Ε, σοσιαλιστές και Δημοκράτες 18, ECR 7, Φιλελεύθεροι 7, η ΓΚΟΕ e 5, η Πράσινη 5, η FDD 3. Μία εγγεγραμμένη πέντε. Παρακαλώ τους συντονιστές να ελέγξουν τα μέλη που ψηφίζουν. Is that done? Every group is in order. Should... Εντάξει, όλες οι ομάδες να προσπαθήσουμε δεύτερη φορά. Άρχεται και πάλι η ψηφοφορία. It's again 74 members, but the... Και πάλι 74 βγαίνουν, 71 μέλη έχει η Επιτροπή μας, όμως τι να κάνουμε. 73, no, it's still too, too much. 73 τώρα, 2 κόμμα παρακαλώ. Όποιος δεν ψηφίζει να βγάλει την κάρτα του από το μηχάνημα για να μην μετράει. Παρακαλώ βγάλτε τις κάρτες όσοι δεν ψηφίζετε. It's not 72, still one too much.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 No, no, it's fine. Κοιτάξτε και τα μέλη του Προεδρείου είναι μέλη των πολιτικών του ομάδων. Πρέπει να τα μετράμε και αυτά. Ωραία. Α ψηφίσουμε τώρα, τα βρήκαμε. No, the people are leaving. I don't know what's going on there. So. Τώρα ψηφίζουν λιγότεροι. 68. Λείπουν τρεις. Πέρα στις φοβερές, σε πάση περίπτωση. Mrs. Έλαβον. Η κυρία Γκριγκούλ 11. Ο κύριος Πλένκοβιτς 46. Ο κύριος Πλένκοβιτς αποδέχεται την εκλογή του. Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για τη τιμή που μου κάνετε. Παρακαλώ, ελάτε στο πρόεδρο. Λοιπόν, έχουμε και ένα σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων για το υπόλοιπο του 14. Έχουμε ακόμα δύο πέμπτες που δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι λίγο ισχνή η παρουσία και είμαι εδώ προκενών εδράνων πέμπτη πρωί, συνήθως αλλά νομίζω για το 14 δεν μπορεί να αλλάξει. Παρακαλώ τη γραμματεία να το φροντίσει με μεγάλη προσοχή για το 15. Να μην έχουμε στην αρχή της εβδομάδα συνεδριάσεις, μετά μια μισή μέρα τίποτα και μετά πέμπτη πρωί. Ε, αυτό κάπως δυσκολεύει το, πρόγραμμά μας. Έχουμε και άλλες δουλειές και έχουμε και εκλογικές περιφέρειες. Γι' αυτό πάντα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν έχεις μια ξεκάρφωτη συνεδρία στην πέμπτη το πρωί να έχεις συχνή παρουσία καλό θα ήταν να το κανονίζαμε διαφορετικά. Εσείς της γραμματείας είστε εδώ όλη μέρα και όλη τη βδομάδα, εμείς έχουμε και κάτι άλλες δουλίτσες. Αυτό δεν καταλαβαίνει η γραμματεία του Κοινοβουλίου, ότι είναι διαφορετικά κάπως τα καθήκοντα των βουλευτών και πρέπει να προγραμματίζεις και τις δραστηριότητές σου. Παρακαλώ να το φροντίσετε. Για το 14 νομίζω αυτό δεν τίθεται πλέον, για το 15 σας παρακαλώ. Συμφωνείτε με αυτό το χρονοδιάγραμμα με αυτές τις προϋποθέσεις. Κατά κανείς. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν ούτως και το χρονοδιάγραμμα. Ερχόμαστε στο σημείο 4. Έγκριση του γλωσσικού προφίλ. Καθεστώς λέει εδώ ρεζίμ. Όταν μιλάς για καθεστώς και γλώσσες αυτό μπορεί να γεννήσει παρεξηγήσεις. Λόγω της σύνθεσης της Επιτροπής μας Νομίζω ότι δεν έχουμε μαλτέζικα, φινλανδικά και ε, γαλλικιανό. Κελτικά. Διαφωνείτε. Βέβαια, όταν αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής θα αλλάζει και το γλωσσικό προφίλ. Αλλά νομίζω αν δεν διαφωνείτε, να αποφασίσουμε ότι εγκρίνεται έτσι το γλωσσικό, γλωσσικό καθεστώς, όπως λέω. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα πριν τις ελληνικές διακοπές θα έχουμε μάλλον συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Ποια μέρα μου λέτε? Την πέμπτη μάλλον. Θα έχουμε και άλλη συνεδρίαση. Όχι. Πέμπτη πρωί. Κατά τα άλλα, η επόμενη τακτική συνεδρίασή μας είναι την 1η Σεπτεμβρίου. Θα παρακαλούσα τους συντονιστές να το σημειώσουν από τώρα. Θα προσπαθήσω την Τετάρτη 9, 9 και 4 να κάνουμε ένα διευρυμένο προεδρείο, αν έχουμε κάπως τακτοποιήσει τα θέματα ε, και έχουν οριμάσει προς απόφαση. Για παράδειγμα, θέλω να το πω και εδώ στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Δεν πρόκειται να μοιράσουμε εκθέσεις τώρα πριν το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει αρκετά γρήγορα να προχωρήσουμε. Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, και προπολογισμό. Αυτά τα θέματα θέλουν ε, γρήγορη αντιμετώπιση και παρακαλώ τι πολιτικέ ομάδε να αρχίσουν ήδη να το σκέφτονται έτσι ώστε την Τετάρτη οι συντονιστέ να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Για να αρχίσουν οι συνάδελφοι πριν από το καλοκαίρι να δουλεύουν τα θέματα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στην επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ προσωπικά και πάλι για την εκλογή. Καλό σας βράδυ.